μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης. Ε, ο εισηγητής έχει το λόγο καταρχήν. Πέντε λεπτά, συνάδελφε Ντάρντεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Εγκρίνοντας την απόφαση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταμορφώνει μια παλιά άτυπη πλατφόρμα δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης σε ένα λειτουργικό και επίσημο δίκτυο συνεργασίας. Είναι σαφές ότι η δημιουργία απασχόλησης είναι αρμοδιότητα όχι των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης. Εξαρτάται από τις πολιτικές απασχόλησης και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Μια πολιτική που έχει βέβαια αποβεί πιο δύσκολη εξαιτία της σημερινή λιτότητας. Όμως οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν ένα σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην ε, τήρηση των στόχων της στρατηγικής 2020 που είναι η αύξηση της απασχόλησης στο 75%. Δεδομένη τη κατάσταση στην Ευρώπη, η οποία αντιμετωπίζει μια ανεργία που μερικέ φορέ φτάνει στο 25% σε χώρε και σε περιφέρειες, κάθε πρωτοβουλία για συντονισμό στον τομέα αυτό πρέπει να προωθείται. Το δίκτυο αυτό λοιπόν θα επιτρέψει πρωτοβουλίες που βασίζονται στη συγκριτική μάθηση, στο bench learning, προκειμένου να μπορούμε να συγκρίνουμε και να εμπλουτιζόμαστε αμοιβαία από την εφαρμογή πολιτικών απασχόλησης ημένα από τους ΔΕ. Πρωτοβουλίες οι οποίες συνεισφέρουν στη μείωση της ανεργίας για όλες τις ηλικιακέ ομάδες και ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες κατηγορίες. Στη μείωση της διάρκειας της ανεργίας για να τα καταπολεμήσουμε τη διαφορετική ανεργία και την κοινωνική τον κοινωνικό αποκλεισμό. Επίσης, το δίκτυο αυτό θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της απασχόλησης, στηρίζοντας στόχους όπως είναι οι πιο ευάλωτες κατηγορίες και θα προωθεί την αξιοπρεπή εργασία, θα βελτιώνει την λειτουργία της αγοράς εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ολοκλήρωσή τη και θα ευνοεί μια γεωγραφική κινητικότητα σε θελοντική βάση και κάτω από ισότιμες συνθήκες για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Το δίκτυο αυτό θα συνεισφέρει επίσης στο να καταγράψει τις αδυναμίες αλλά και τα προσόντα των ε, ατόμων που ζητούν απασχόληση και των ε, εργοδοτών. Θα διαπιστώσετε λοιπόν ότι οι στόχοι του δικτύου αυτού είναι φιλόδοξοι. Έχει ρόλο να αναλύσει, να κάνει ανταλλαγέ, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να κάνει προτάσεις στον τομέα των πολιτικών απασχόλησης. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί πρέπει όλες οι χώρες μέλη να συνεργαστούν με τους άλλους φορείς που δρούν στο, στην αγορά εργασίας. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται η παρουσία όλων γύρω από το ίδιο τραπέζι για να μπορέσουν να γίνουν επιτυχείς συζητήσεις. Τι ερμηνεία πρέπει να δώσουμε στο κείμενο της νομικής βάσης για την υποχρεωτική ή τη θελοντική βάση του δικτύου αυτού. Από τις συζητήσεις που κάναμε δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε γιατί υπάρχουν ερμηνείες αντιφατικές ανάμεσα στο Συμβούλιο από τη μια και την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο από την άλλη. Το Συμβούλιο θέλει να προσθέσει μονομερή δήλωση που να διευκρινίζει την ερμηνεία που δίνει για εθελοντική βάση συμμετοχής όλων. Η Επιτροπή Απασχόληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτείνει επίση να προσθεθεί στη συμφωνία αυτή μια άλλη δήλωση χωρί να αμφισβητεί την ερμηνεία. Δηλαδή να υπάρξει συμμετοχή όλων υποχρεωτικά. Γιατί αυτό μόνο διασφαλίζει μια ισότιμη εφαρμογή. Ακόμα ομω και με τη διαδικασία αυτή καταλήγουμε σε ένα κείμενο τελικά χωρί γωνίε. Δεν ενισχύει αυτό όμω την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων στα πλαίσια τη συναπόφαση. Χρειάζεται επίσης καλή συνεργασία στο δίκτυο. Το δίκτυο πρέπει να συνεργάζεται με τους κοινωνικούς εταίρους, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, αλλά και τις υπηρεσίες απασχόλησης με όλους τους φορείς. Χρειάζεται επίσης συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι της γραμματείας που διασφαλίζει η Επιτροπή και την Επιτροπή Απασχόλησης ΕΜΚΟ η οποία έχει καθεστώς παρατηρητή που όμως μερικές φορές ε, οι συνεδριάσεις γίνονται σε περιορισμένη σύνθεση. Προσπαθήσαμε με την απόφαση αυτή η οποία θέλει συνεργασία μεταξύ όλων των εταίρων, θέλει επίσης και την εφαρμογή δραστηριοτήτων του δικτύου σε χώρες όπου έχουν αρμοδιότητες που ρυθμίζονται στο εσωτερικό της χώρας μεταξύ διαφορετικών ε, θεσμών όπως το Βέλγιο. Η συμφωνία αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι, απορρέει από μια καλή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα γίνει πράξη με τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας και παρά τις αποκλήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, άλλους ε, εισηγητές και την πρόεδρο Περβένς ε, Μπερές, της οποίας η εμπειρία και η επιμονή είναι δεδομένα. Για να καταλήξω, το νέο αυτό εργαλείο Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής θα δώσει μια νέα όθηση στην καταπολέμηση της ανεργίας, ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων και στην καταπολέμηση των κοινωνικών αποκλεισμών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε Ντάρντεν και τώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Επίτροπος Άντορ. Πρόεδρε, Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, καταρχά να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Νταρντά και του σκιώδει εισηγητέ για το έργο του, προκειμένου να παρατωθεί το νομοθετικό έργο για την απόφαση αυτή για τι δημόσιε υπηρεσίε απασχόληση. Η έγκριση τη απόφαση αυτή ήταν ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και δίκτυα για να καταπολεμήσει την ανεργία. Η απόφαση αυτή θα βελτιώσει τη λειτουργία των δημόσιων αυτών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θα στηρίξει έτσι περαιτέρω ε, τον συντονισμό των ε, πολιτικών απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δημόσιε αυτέ υπηρεσίε βρίσκονται στην πρώτη γραμμή τη αντιμετώπιση τη ανεργία και προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην εσωτερική αγορά. Έχουν πολύ διαφορετικά επίπεδα επιδόσεων, ωστόσο, ακόμα και κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2013, οκτώ κράτη-μέλη έλαβαν ε, αναχώρα συστάσεις για τις δικές τους δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. Κατά πάσα πιθανότητα θα ξανασυμβεί αυτό στο Ευρωπαϊκό Εξάμενο 2014. Επιπλέον, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης είναι φορείς καθοριστική για την εφαρμογή των ε, συστάσεων του Συμβουλίου για τη δημιουργία της εγγύησης των νέων. Η δημιουργία και η χρήση του ταμείου αυτού ε, είναι κάτι που θα πρέπει να ε, το χειριστούν οι υπηρεσίες για την ανεργία, για τους ανέργους στις επιμέρους ε, θα πρέπει λοιπόν να αναλυθούν συγκεκριμένε πρωτοβουλίε όπω ένα κοινό σύστημα αναφορά που να βασίζεται σε αποδικά στοιχεία με συγκριτική αξιολόγηση και αμοιβαία εκπαίδευση με την αμοιβαία ε, συνδρομή μεταξύ των μελών του δικτύου και την υλοποίηση στρατηγικών δράσεων για τον εξυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών απασχόληση. Αυτά θα πρέπει να βοηθήσουν τα κατημέλη και τι υπηρεσίε του, να αυξήσουν το επίπεδο των επιδόσεών του και να προσφέρουν ε, επιλογέ του σε εργασία. Ξέρω ότι το Συμβούλιο σκοπεύει να γκρίνει μονομερή δήλωση, τονίζοντα την οικειοθελή συμμετοχή των κατών σε αυτό το δίκτυο και ε, δηλώνοντα ότι θα συμμετέχουν παρόλα αυτά όλα τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταστήσει σαφέ σε ε, πολλέ ευκαιρίε ότι δεν συμμερίζεται αυτή τη νομική ερμηνεία. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη στιγμή τη έγκριση του νομοθετήματο στο Συμβούλιο θα δημοσιεύσει επίση δήλωση εκφράζοντα την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη σαφήνεια για την ερμηνεία τη νομική βάση. Καταλαβαίνω ότι το σώμα σα θέλει να κάνει κάτι ανάλογο με μία δήλωση. Γιατί είναι σημαντικό να υπάρξει νομική ασφάλεια εδώ. Διότι αυτό που προέχει σήμερα είναι να εγκριθεί η απόφαση. Να εγκριθεί η απόφαση και να είμαστε βέβαιοι ότι θα υλοποιηθεί. Αυτό μετράει για του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αναζητούντε εργασία και οι εργοδότε το ίδιο ε, ανησυχούν για το να έχουν καλέ δημόσιε υπηρεσίε μεταξύ των οποίων ε, υψηλή ποιότητα ε, προσφορά από τι δημόσιε υπηρεσίε απασχόληση. Καλώ λοιπόν εσά, τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, να εγκρίνετε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε Άντορ. Και τώρα οι αγορητέ ε, εξ των πολιτικών ομάδων, ο κύριος Μπέκαρ για δύο λεπτά. Αξιότιμα κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, αποτελεσματική και επικοδομητική συνεργασία μας. Μαζί του ε, μπορέσαμε Ε, ως ΕΛΚ να πραγματοποιήσουμε με επιτυχία την πρόταση της Επιτροπής. Μπορέσαμε στις τριμερείς, ε, ε, στον τριμερή διάλογο να κάνουμε καλές συζητήσεις. Έχουμε τώρα καλό μέσον στην πάλι κατά της ανεργίας και ήδη στη φάση της πρόληψης έχουμε σημειώσει επιτυχία. Αυτό είναι σημαντικό πρόσθετο βήμα. Ε, χαίρομαι πολύ με αυτή την έννοια της, του bench learning, συγκριτική μάθηση. Ε, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μαθαίνουν το ένα από το άλλο. Επιτυχή μοντέλα όπως ε, ε, το αυστριακό πρόγραμμα για την εγγύηση για την νεολαία θα πρέπει να βρουν μιμητές και η Αυστρία μπορεί να μάθει από άλλους από τις σκανδιναβικές χώρες για παράδειγμα που στοχευμένα φροντίζουν οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι να παραμείνουν στην θέση εργασία τους και να μην ε, ε, εξαναγκαστούν να αποχωρήσουν πρόωρα. Είναι σημαντικό για το δίκτυο των ε, ευρωπαϊκών διοικήσεων, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια τα οποία είναι σημαντικά και για την συνέχεια του bench learning. Ε, έτσι θα μπορούν με μεγαλύτερη ακρίβεια να αξιολογούν τις επιτυχίες άλλων χωρών. Είναι επίσης θετικό το γεγονός ότι το ε, EURES, η Ευρωπαϊκή Ελεκτρονική Διεύθυνση, η πύλη αυτή έχει ε, θα ενισχυθεί και θα γίνει ευρύτερα γνωστή. Ε, ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο συνάδελφος Κοστέλο για 1,5 λεπτό. Κύριε, ε, κύριε Κοστέλο, ευχαριστώ Πρόεδρε να επενέσω τον κύριο Νταρντέν για την εργασία του επί της έκθεσης αυτής για τον απλό λόγο ότι έχουμε 26 εκατομμύρια που είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη συμπεριλαμβανομένων των 100.000 ε, στη δική μου την εκλογική περιφέρεια και μόνον. Αυτό σημαίνει επειδή δεν υπάρχουν αρκετέ θέσει εργασία και ο τρόπο να αντιμετωπίσουμε την ενεργεία είναι η Ευρώπη επιτέλου να στρέψει την προσοχή τη από τη λιτότητα προ την βιώσιμη ανάπτυξη. Και ταυτόχρονα η στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των δημόσιων δημόσιων υπηρεσιών του απασχόληση είναι κάτι που θα διαρματίσει σοβαρότατο ρόλο. Η Ευρώπη ε, θα πρέπει να έχει τέτοιε δημόσιε υπηρεσίε που να λειτουργούν καλύτερα, αποτελεσματικότερα και να συνεργάζονται μεταξύ του. Θα πρέπει να στηρίξουμε μεν του δε, ιδίω κατά την υλοποίηση τη εγγύηση ε, για του νέου, για την νεολαία. Θα πρέπει καλύτερε τέτοιε δημόσιε υπηρεσίε να μα επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα προβλήματα τη κοινή αγορά και τη ανεργία και να αντιποκριθούμε με αποτελεσματικότητα. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων με κυβερνητικών ε, οργανώσεων, των ε, δημόσιων φορέων και των αρχών τοπική αυτοδιοίκηση ώστε να μπορέσουν οι άνεργοι να ανακάμψουν και να βρουν δουλειά. Θα πρέπει να φροντίσουμε οι επενδύσει που προέρχονται και τα κονδύλια που προέρχονται από το Κοινωνικό Ταμείο λόγω Χάρη αλλά και άλλα ταμεία να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στην Ιρλανδία. Υπάρχει μια σοβαρότατη μεταρρύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόληση με νέου κανόνε να επιβάλλονται και με πρόσωπα που επιτέλου να μπορούν να απευθυνθούν σε τέτοιε υπηρεσίε και να βρουν σιγά σιγά το δρόμο του προ την αγορά απασχόληση. Επιτέλου, η Ιρλανδία θα πάρει μέρο σε αυτή την πρωτοβουλία και γι' αυτό στηρίζω την πρόταση όλε οι χώρε να συμμετάσχουν στο δίκτυο αυτό. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κοστέλο. Ο κύριος Μπένιον, δυόμιση λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η απόφαση αναγνωρίζει τη σημασία της πανευρωπαϊκής συνεργασίας στην απασχόληση. Ιδιαίτερα τώρα που η ανεργία έφτασε σε ύψη ρεκόρ σε κάποια κράτη-μέλη και κάποια τμήματα του πληθυσμού ε, έχουν ε, πεταχτεί έξω από την αγορά εργασίας. Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόληση αντιμετωπίζουν μεγάλες πιέσεις, κοινέ καμιά φορά στην Ευρώπη. Το δίκτυο θα τους δώσει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών θα ενισχύσει το υφιστάμενο δίκτυο και θα αυξήσει τη συνεργασία και με άλλους εμπλεκομένους ε, όπως μη κυβερνητικέ και το Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό όταν πρόκειται για την εφαρμογή πρωτοβουλειών όπως η εγγύηση για την νεολαία. Και το bench learning, η συγκριτική μάθηση θα βελτιώσει τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών απασχόληση γιατί θα εντοπίσει πού πάνε καλά και θα μπορούν κι άλλοι να μάθουν από αυτή τη διαδικασία. Το δίκτυο θα στηρίξει πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνήμα των νέων που δεν βρίσκονται σε απασχόληση ή εκπαίδευση ε, και ε, λέγονται νίτς για να, στη, να, μπουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Το τελικό κείμενο αναφέρεται σε αντιστοιχεία και ελλείψεις δεξιοτήτων. Ο εντοπισμός των ε, ελλείψεων δεξιοτήτων πρέπει να είναι προτεραιότητα, ούτω ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι καλύπτουμε όλους τους ε, πολίτες, όχι μόνο τους νέους, με τις δεξιότητες που χρειάζεται για να εργαστούν στην ε, αγορά εργασίας. Αυτό το δίκτυο θα μας βοηθήσει σε όλη την Ένωση. Επίσης θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε την κάλυψη θέσεων εργασίας από εκείνους που αναζητούν απασχόληση και θα αυξηθεί και η κινητικότητα. Η συνεργασία που διευκολύνεται από το δίκτυο θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του 2020 για έξυπνη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια πολύ θετική απόφαση και καλό όλα τα κράτη-μέλη να την υπερψηφίσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπένιον. Και τώρα η κυρία Λάμπερτ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του. Είναι αλήθεια ότι όταν κοιτάμε τα θέματα σχετικά με την ανεργία, τίθεται το ζήτημα της ποιότητας, τι ενημέρωση έχουμε από τη διοίκηση και διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ σημαντικά στοιχεία αυτά γιατί επηρεάζουν την ζωή των ανθρώπων. Πρέπει να θυμόμαστε ότι για να υπάρχει πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου δημόσιε υπηρεσίες πρέπει να υπάρχει μια ατζέντα συμμετοχή για όλου. Φυσικά και πρέπει να μαθαίνουμε μένα από του δε, να ανταλλάσσουμε εμπειρίε. Εποφελούμαστε από αυτό. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η συμμετοχή όλων των χωρών μελών είναι κάτι πολύ σημαντικό και ειλικρινά πιστεύω ότι τα επιχειρήματα που ακούμε κατέληξαν στο να δυσκολέψουν κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι κοινή λογική. Φυσικά και πρέπει να ανταλλάσσουμε εμπειρίε, να προσφέρουμε ευκαιρίες για εμπειρίε τους ανθρώπους και αυτό γίνεται με την εγγύηση για τους νέους, για την απασχόληση. Πρέπει να αντιμετωπιστεί μακροχρόνια ανεργία και κυρίως να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες. Η συνεργασία με όλους τους φορείς είναι κάτι που όλοι πιστεύουμε πως θα προσθέσει στο δίκτυο. Και όχι μόνο με τις υπηρεσίες απασχόλησης τις περιφερειακές και τις τοπικές, αλλά και όλους τους φορείς που εκπροσωπούν τους άνεργους και τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους. Ελπίζω τέλος πάντων να ξεπεράσουμε αυτά τα αρχικά εμπόδια και να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο να είναι ιδιαίτερα επικοδομητικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Λάμπερτ. Ο συνάδελφος Καμπρνόχ δεν είναι εδώ, οπότε ο κύριο... Κυρία Ζούμπερ. Ευχαριστώ. Είναι σαφέ ότι το πρόβλημα τη ανεργία είναι κεντρική σημασία και αφορά πάρα πολλού πολίτε και κυρίω νέου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω η επίλυση του προβλήματο θα πρέπει να περάσει κυρίω από τι επενδύσει, ιδίω στι χώρε των οποίων η παραγωγή, η τεχνολογία και η έρευνα, η ανάπτυξή του δεν είναι αρκετέ. Εκεί υπάρχουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργία. Θα πρέπει λοιπόν να αναλυθούν τέτοια μέτρα ώστε να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση και να μην καταστρέφονται αντιθέτω οι θέσει εργασία. Θα πρέπει να κοιτάξουμε ότι έχουμε δημιουργήσει κατακαιρματισμένε επιμέρου αγορέ και υποφελούνται από την εσωτερική αγορά άλλε χώρε περισσότερο από ότι κάποιε. Ε, οπότε εδώ πρέπει να αναζητήσουμε και μια εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται στι χώρε του με σεβασμό και να κοιτάξουμε να μην δημιουργηθεί ένας, μια ομάδα των ισχυρότερων οικονομικά χωρών και των χωρών που θα εξάγουν φθηνό εργατικό δυναμικό. Θέλουμε ε, να ληφθούν υπόψη οι προτάσει που ε, υποβάλαμε, ιδίω αυτέ για τη δικτύωση των συνεκλειστικών οργανώσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ συνάδελφε Τζούμπερ. Και τώρα 1,5 λεπτό η κυρία Ισαγιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η συνεργασία των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα με δεδομένη την κατάσταση της απασχόλησης στην Ευρώπη σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι η απασχόληση και η κοινωνική ασφάλιση οργανώνονται με διαφορετικό τρόπο στα διάφορα κράτη-μέλη και είναι θέμα κρατών μελών. Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι σε βάση εθελοντική με ανταλλαγή εμπειριών και είμαι βεβαία ότι θα μπορέσουμε έτσι να επιτελέσουμε πρόοδο. Όπως είπε και ο Επίτροπος, η Ευρωπαϊκή Εγγύηση για την Νεολαία και η εφαρμογή της ε, συνεπάγεται βελτίωση σε πολλά κράτη-μέλη. Η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης είναι σημαντική ε, για την απασχόληση των νέων και θέλω να αναφέρω και τις δυνατότητες ε, να βρουν απασχόληση και άνθρωποι με αναπηρίες. Νομίζω ότι αυτές οι ομάδες χρειάζονται μια βοήθεια για την εξέβρεση απασχόλησης Οπότε καλό θα ήταν να προσέξουμε περισσότερο ε, μέσω των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης το ζήτημα της απασχόλησης για άτομα με αναπηρίες. Είναι πολλοί οι άνθρωποι με αναπηρίες που είναι άνεργοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα η κυρία Ρέγνερ 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω με αυτή την ε, ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά και για πολλά άλλα θέματα. Πάνω από 26 εκατομμύρια άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες είναι άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι καταστροφικά τα στοιχεία για τους νέους. Υπάρχουν ε, χώρες όπου το 50% των νέων είναι άνεργοι. Ε, πρόκειται για μια καταστροφή που δεν πρέπει να κουραζόμεθα να προβάλλουμε. Πώς μπορούμε να την καταπολεμήσουμε αυτή την ανεργία, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, πώς μπορούμε να ξαναφέρουμε τον κόσμο στην απασχόληση. Βέβαια, η... χρειαζόμαστε κυρίως μεγάλες μακροοικονομικές λύσεις που ως σοσιαλδημοκράτες πάντοτε τις προωθούμε ε, να εγκαταλείψουμε τη λιτότητα και να πάμε σε αύξηση των επενδύσεων, εγγύηση των, για την νεολαία. Πρέπει όμως να δούμε και τις μικρές βελτιώσεις, ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών ευρέσεως εργασίας. Είναι σημαντικό αυτό. Ε, βέβαια, ε, δεν θα λυθεί έτσι η μαζική ανεργία, αλλά η καλύτερη συνεργασία των ε, υπηρεσιών απασχόλησης μπορεί να ε, απλούς, να, να, να βοηθήσει ανθρώπους να βρουν εργασία. Όλοι ε, αξίζουν μια τέτοια ευκαιρία. Ε, οι εργοδότες, οι, τα συνδικάτα θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται όπως και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και βεβαίως το σύστημα πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε Ρέγνερ. Και τώρα για 1,5 λεπτό η κυρία Γιασλοβιέτσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σαν στόχο να επισημοποιήσει τη συνεργασία μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης, δημιουργώντας ένα δίκτυο. Αξίζει το κόπο να τη στηρίξετε, γιατί το θέλει είναι πολλά. Δημιουργείται έτσι μια πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Οι χώρες μέλη έχουν διαφοροποιημένα μοντέλα και συστήματα δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης. Διαθέτουν διαφορετικά εργαλεία, διαφορετικά μέσα και διαφορετικά πλαίσια μέσα στα οποία λειτουργούν. Και γι' αυτό μέχρι τώρα ήταν αδύνατον να φτιάξουμε μια πραγματική αγορά εργασίας. Θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε διαφορετικά μοντέλα διαφορετική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης χάρη σε αυτό το δίκτυο. Θα μάθουμε από τα λάθη των άλλων. Μπορούμε έτσι να επιλέξουμε τις λύσεις οι οποίες έχουν αποδειχθεί ορθές. Μια τέτοια πλατφόρμα συνεργασίας θα ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση. Βέβαια δεν υπάρχει πλατφόρμα συνεργασίας μέσα στην οποία να συμπεριλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες. Μια τέτοια πρόταση όμως βοηθάει στο να καταλήξουμε σε καλύτερη συνοχή της αγοράς εργασίας μεταξύ των χωρών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κυρία ε, Γιασλοβιέσκα. Για ένα λεπτό κύριο Σκοφεράτη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είναι γνωστό ότι περισσότερε θέσει απασχόληση μπορούμε να έχουμε μόνο με αναπτυξιακέ πολιτικέ. Και τέτοιε αναπτυξιακέ πολιτικέ μπορούμε να έχουμε μόνο με κρατικέ επενδύσει, ώστε να τονωθούν οι ιδιωτικέ επενδύσει και να υπάρχει ανταγωνιστικότητα στι επιμέρου απερχίε. Όμω είναι εξίσου προφανέ ότι όλα αυτά που εξυπηρετούν για να γίνει πιο αρμονική και εύρυθμη λειτουργία τη ε, αγορά απασχόληση, για να εξισορροπηθούν η ζήτηση και η προσφορά και να αρθούν οι φραγμοί που παρουσιάζονται στην ε, πρόσβαση τη ε, αγορά εργασία των νεωτέρων, όλα αυτά τα έλεγα μπορεί να είναι πολύ σημαντικά παράπλευρα αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν, μάλλον είναι προποθέσει. Γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει τι δημόσιε υπηρεσίε απασχόληση να τι δούμε ω πυλώνε αυτή της προσπάθειας. Θα πρέπει να προωθηθούν ώστε να είναι σαφέ για όλου περί τίνο πρόκειται και τι δεσμοί, τι συσχετισμοί πρέπει να δημιουργηθούν. Ο δρόμο αυτό πάντω είναι σαφώ σωστό και πρέπει να τον επιδιώξουμε με τόλμη. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κοφεράτη. Κύριο Κράουλη, στα πλαίσια της διαδικασίας Catch the Eye. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για την ανεργία και τις λύσεις. Πολλές φορές ξεχνάμε ότι η ανεργία δεν προκαλείται τόσο από το κράτος, αλλά από η, απασχόληση δεν προκαλείται από το κράτος, αλλά από τις επιχειρήσεις. Δράση λοιπόν θα πρέπει να ε, αναλυθεί σε αυτά τα επίπεδα, ούτω ώστε να δώσουμε στον κόσμο ε, δεξιότητες και δυνατότητες απασχόλησης, αλλά να διασφαλίσουμε ότι η εκπαίδευση, οι δεξιότητες θα είναι κάποιο επίπεδου. Ε, αν δώσεις ψάρι σε κάποιον, ε, του δίνεις τροφή για μία μέρα, αν του μάθεις να ψαρεύει, τον ταΐζεις για μια ζωή. Αυτό είναι σημαντικό και με την ανεργία των νέων, να δώσουμε δεξιότητες στον κόσμο, να διασφαλίσουμε ότι έχουν τις δεξιότητες για τις καινούργιες θέσεις εργασίας. Ε, όχι να ε, κάνουμε ε, εκπαίδευση ή ε, σεμινάρια μετάβασης, αλλά να είναι πραγματικές παρεμβάσεις αυτές στην αγορά εργασίας και την απασχόληση. Ευχαριστώ πολύ. Και έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία Catch the Eye και δίνω το λόγο στον Επίτροπο Άντορ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή κ. Ντάρντεν για τη συμβολή του για την επίτευξη συμφωνίας με το Συμβούλιο για την απόφαση για τις δημόσιες υπηρεσίες. Τα μέλη συζήτησαν την πρόταση σήμερα στα πλαίσια και με φόντο την υψηλή ανεργία στην Ευρώπη. Όμως ε, το θέμα σήμερα είναι ότι όχι μόνο έχουμε υψηλή ανεργία, αλλά ότι είναι πολύ διαφορετική η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλωμένη καμιά φορά εις ό,τι αφορά το τομέα της απασχόλησης. Όταν ε, πηγαίνουμε στην Αυστρία ή τη Βαβαρία, που ήμουν εκεί την Κυριακή, ε, ε, σκεφτόμαστε ότι κάτι πηγαίνει πάρα πολύ καλά στις χώρες αυτές σε ό,τι αφορά την απασχόληση. Και οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης είναι μέρος της απάντησης. Από την άλλη πλευρά, σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, Υπάρχουν τεράστια προβλήματα ακόμα και σήμερα. Όχι μόνο αδυναμίες των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης, αλλά ε, υπάρχει μια συνθετότητα ε, ε, προβλημάτων. Δεν υπάρχει χρυσή λύση για να λύσουμε την, ε, το πρόβλημα της ανεργίας. Βεβαίως και θα πρέπει να βελτιωθούν οι μακροοικονομικές συνθήκες και πρέπει να βρούμε λύση για την αύξηση των επενδύσεων. Αλλά θα πρέπει να ε, κάνουμε πιο λειτουργική και την αγορά εργασίας. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι και οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης πιο αποτελεσματικές. Το νέο δίκτυο των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης θα βοηθήσει να αυξηθεί η, η απόδοση αυτών των υπηρεσιών με αμοιβαία μάθηση και τεχ, προγράμματα τεχνικής υποστήριξης. Η πολιτική σημασία αυτού του δικτύου ε, πάει πολύ πιο πέρα. Πριν από δύο χρόνια στο, στη δέσμη μέτρων απασχόλησης ε, ε, για να αντιμετωπίσουμε την ύφεση παρουσιάσαμε το όραμα της Ευρωπαϊκής Αγοράς Εργασίας και πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ε, βρίσκουν λύσεις στην ανεργία ε, πηγαίνοντας να εργαστούν στο εξωτερικό. Ε, εδώ χρειάζεται βέβαια να υπάρχουν γλωσσικές δεξιότητες για να αυξηθεί η κινητικότητα και πρέπει να βοηθήσουμε εκείνους που θέλουν να αξιοποιήσουν την ελευθερία διακίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως θα ήταν λάθος να υποθέσουμε ότι η πρόταση αυτή αφορά μόνο την κινητικότητα της εργασίας η εφαρμογή σημαντικών δεσμεύσεων όπως η εγγύηση για την νεολαία εξαρτάται, εξαρτώνται και από λειτουργικότερες, αποτελεσματικότερες δημόσιες υπηρεσίες απασχόληση σε πολλά κράτη-μέλη. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η σημερινή πρόταση και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να υπερψηφιστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε Άντορ. Και τέλος, ο εισηγητής για ένα λεπτό, ο κύριος Ντάρντεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ανάγκη να καταπολεμήσουμε με όλα τα δυνατά μέτρα συντονισμένα την ανεργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να έχουμε γρήγορη εφαρμογή τη εγγύηση για του νέου είναι κάτι το προφανέ και το θύμισαν όλοι σε αυτή τη συζήτηση. Να ευχαριστήσω όλου του παρεμβαίνοντε για τη στήριξή του. Σε ό,τι αφορά τι τροπολογίε που υποβλήθηκαν για την ψηφοφορία, εγώ θα έλεγα να μην τι στηρίξουμε, διότι το πνεύμα τη έκθεση θα αλλοιωθεί ε, και το ίδιο και συμβαστικέ λύσει αν ψηφίσουν οι τροπολογίε συμφωνία με το Συμβούλιο. Θα συμφωνήσουμε με τον Επίτροπο ότι τα μέτρα πρέπει να ε, εγκριθούν σε αυτήν την θητεία, ώστε το δίκτυο να μπορέσει να αρχίσει να λειτουργεί αμέσω, όσο το δυνατόν συντομότερα, με πλήρη τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε Ντέρντεν. Ε, ολοκληρώσαμε τη συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στι 6 ε, και διακόπτουμε μέχρι την έναρξη τη ψηφοφορία ψηφοφορίας στις 6. Thank you. Thank you.